Λίμπε έχει ζητήσει διόρθωση για το άρθρο του κανονισμού βάσει το άρθρο 351 του κανονισμού στο τέταρτο εδάφιο. Οι αλλαγές έχουν, θα θεωρηθούν εγκεκριμένες εάν μέσα σε ένα 24ωρο ε, ένας βουλευτής ε, ή ομάδα βουλευτών που να φτάνουν τον ε, κατάλληλο αριθμό ψήφων δεν προβάλλουν αντίρρηση. Ο τίτλος θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της τρέχουσα συνόδου.